εκτός της παρεμβάσης τους, αρκεί να μην ξεπερνούν τις 200 λέξεις. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης, τη συζήτηση για τη Μαυριτανία και κυρίως την περίπτωση του Μπιράμ Νταχ Αμπέιντ. Το λόγο έχει πρώτα η κυρία Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Μαυριτανία επίσημα κατηρίγησε την σκλαβιά από το 1981. Στην πρακτική όμως η ε, δουλεία εξακολουθεί να υπάρχει. Ε, μη κρατικέ οργανώσεις ε, όπως η αλλά και άλλες SOS Clubs αναφέρουν συνεχώς αυτές τις περιπτώσεις δουλείας. Η κυβέρνηση της Μαυριτανίας καλά θα έκανε λοιπόν να λάβει σοβαρά υπόψη στην την εργασία αυτών των οργανώσεων και μάλιστα να τις αντιμετωπίσει και ως υποστήριξη στον αγώνα για την εξάλληψη της δουλείας. Όμως η κατάσταση δείχνει ακριβώς το ίδιο. Σήμερα λοιπόν εμείς με το ψήφισμά μας καλούμε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα ε, και να μην διώκει πλέον τους ε, ε, πολιτικούς ακτιβιστές. Θέλουμε να απελευθερωθούν όσοι έχουν συλληφθεί. Πρώτα απ' όλους ο κύριος Μπιράμτα Αμπάιτ. Στη Μαυρτανία, εάν πραγματικά επιθυμούμε να εξαλείψουμε τη δουλεία, τότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη φτώχεια αυτών των ανθρώπων. Η ομάδα των χαρατίν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει γη. Γη στην οποία βρίσκονται και εργάζονται εδώ και αιώνε, γη την οποία καλλιεργούν. Η κυβέρνηση τη Μαυριτανίας καλείται λοιπόν να δραστηριοποιηθεί σοβαρά. Και οι διεθνεί επιχειρήσει οι οποίε δραστηριοποιούνται στη Μαυριτανία καλούνται και αυτέ να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει εξαναγκαστική και μάλιστα παιδική εργασία. Είναι και καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσει και αυτή ότι στις εμπορικές σχέσεις με τη Μαυριτανία ούτε και έμεσα δεν θα γίνεται ανεκτή η δουλεία και η σχετική εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση για την ε, ε, Μαυριτανία και τον Μπιράμ Μπέιτ δεν είναι κάτι εύκολο για μένα. Εγώ πρότεινα το ζήτημα αυτό ε, με τη διαφορά άλλων θεμάτων που έχουμε συζητήσει εδώ, πρέπει να πω ότι επανειλημμένα έχω συναντήσει τον Μπιράμ Ντάν Αμπέη, ακτιβιστή ε, για το θέμα της ε, κατάργησης της δουλείας. Ε, συζητούμε το θέμα αυτό εδώ και ζητώ επομένως με σαφήνεια από τις μαυρετανικές αρχές να ελευθερώσει τον άνθρωπο αυτό ο οποίος παλεύει για το καλό της χώρας του. Θα πρέπει η Μαυριτανία να βγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο της άρνησης της πραγματικότητας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και να να αφομοιώσει ε, τα δεινά της ε, ε, δουλείας έτσι ώστε να επιτρέψει την επιβίωση του λαού της Μαυριτανίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζιβενάσκα. Ευχαριστώ πολύ. Παρότι λοιπόν είμαστε ήδη στο 2014, έχουμε εδώ μια χώρα όπου βλέπουμε τη σύγχρονη δουλεία γιατί στη Μαυριτανία ζουν πραγματικοί σκλάβοι. Έχουμε τα αφεντικά που αποφασίζουν για τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Εγώ λοιπόν ε, καταδικάζω απερίφραστα τέτοιου είδους ε, καταστάσεις ε, οι οποίες απαγορεύονται και από το Σύνταγμα της ίδιας της χώρας. Καλώ λοιπόν την κυβέρνηση της Μαυριτανίας να απελευθερώσει πάρα αυτά τον κύριο Μπιράμ Νταχ Αμπέιτ, ακτιβιστή γιατί αν δεν αφαιθεί ελεύθερος αυτό θα είναι ένας κόλαφος για τον αγώνα κατά της ε, δουλείας. Ε, πρέπει λοιπόν να σας πω ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να δεχόμεθα τα οικονομικά συμφέροντα. Ε, ορισμένοι εξημών ε, τα τελευταία χρόνια είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ε, Μπιράμντα Αμπέιτ, ε, ο οποίος είναι κατά της ε, δουλείας, που δυστυχώς όμως η δουλεία εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα του. Είναι ο γιος πρώην σκλάβων και ο άνθρωπος αυτός τάσεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι μόνο στην διεθνή σκηνή αλλά και κυρίως στην πατρίδα του στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που επιθυμεί να ενημερώσει τους συμπολίτε του αλλά συνελήφθη και ο ίδιος και πολλοί άλλοι συμπολίτε του κατηγορείται λοιπόν και ενδεχομένως υπάρχει την πιθανότητα να καταδικαστεί και σε θάνατο. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθούν όλοι οι άνθρωποι αυτοί ελεύθεροι και η Μαυριτανία να ε, τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει μέσω διεθνών συνθήκων. Ελπίζω λοιπόν αυτό το ψήφισμα να βοηθήσει να ξεκινήσει ο διάλογος με την κυβέρνηση της Μαυριτανίας για να αρθούν πλέον τέτοιου είδου καταστάσει. Ευχαριστώ κύριο Σκοράου. Σύμφωνα με τελευταίο η ε, ε, τελευταία έκθεση ε, των Ηνωμένων Εθνών είναι πάνω από το 40% του πληθυσμού που υποχρεώνεται να ζει κάτω από έναν αφέντη. Αυτή είναι η φοβερή αλήθεια. Υπάρχουν και άλλες μορφές παραβίασης σχετικά με την απλήρωτη εργασία, σχετικά με την, εργασία, την παιδική εργασία, σχετικά με παιδιά τα οποία γεννιούνται σκλάβοι. Υπάρχει ακόμα στην η κατάσταση του να γεννιέται κανείς σκλάβος και να είναι ιδιοκτησία ε, του ε, αφεντικού. Ε, κάθε μέρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ζουν χωρίς δικαιώματα. Τον προηγούμενο χρόνο πάρα πολλοί ακτιβιστές έχουν φυλακιστεί και μεταξύ των οποίων και ο Μπιράν Ντάχα Αρμπάιντ του οποίου το μόνο έγκλημα ήταν να καταδικάζει και να αγωνίζεται κατά της δουλείας. Ζητάμε λοιπόν την άμεση απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων για λόγους συνείδησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στεπρέ. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος ε, των φιλελευθέρων θα ήθελα δημόσια να εκφράσω την στήριξή μας ε, σε τούτο το ψήφισμα ε, που ζητά άμεση απελευθέρωση του Μπιράμ Ντάχ Αμπέιτ καθώς επίσης και των άλλων ακτιβιστών και που καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή δουλείας. Όμως, ε, λυπάμαι γιατί οι δύο μεγάλες ομάδες δεν δέχτηκαν παραγράφους που ζητήσαμε. Είχαμε ζητήσει ε, ε, να αναφέρεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, η κυβέρνηση της Μαυριτανίας να προσυπογράψει την, το τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διαφρικανικής διάσκεψης. Επίσης ζητήσαμε να γίνει αναφορά στο άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού. Ούτε αυτό έγινε. Επίσης είχαμε ζητήσει να ξεκινήσει διαδικασίες η Κομισιόν βάσει του άρθρου 96 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό ε, δεν έγινε ε, δεκτό. Ε, στη διάρκεια των συζητήσεων ακούσαμε ότι για λόγους ισορροπίας δυνάμεων δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν αυτά τα στοιχεία και αυτό πραγματικά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Η κυρία Σένερα Ροδρίγκες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το άρθρο 4 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μάλιστα πριν από λίγο εορτάσαμε, απαγορεύει κάθε μορφή δουλείας και σήμερα, 66 χρόνια μετά, 21 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο είναι θύματα εξαναγκαστικής εργασίας. 4,5 εκατομμύρια ε, καταναγκαστικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Θα πρέπει να στυλιστεύσουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ε, που εφαρμόζονται και που συνιστούν απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το άρθρο 4 της Οικουμενικής Διακήρυξης σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να θελοτυφλούμε ή να κάνουμε τα στραβά μάτια θα πρέπει να απαιτήσουμε από τη Μαυριτανία να απελευθερώσει αμέσως τον Πυράμ Ντάχ Αμπέιτ και να καταργήσει και εμπράκτος τη δουλεία. Επίσης να λάβει μέτρα ώστε τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμποδίσουν, να υποχρεώνουν μάλλον τις πολυεθνικές να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες ότι η Μαυριτανία ήταν η τελευταία χώρα στον κόσμο που κατήργησε τη δουλεία το 1981. Και μόνο αργότερα ποινικοποιήθηκε η δουλεία. Βέβαια, παρά την ποινικοποίηση, έκτοτε είχαμε ελάχιστες διώξεις για το αδίκημα του εξανδραποδισμού. Η Μαυριτανία μάλιστα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, τουλάχιστον 4% που υφίστανται κάποια μορφή σύγχρονης δουλείας. Δείχνουν λοιπόν όλα τα στοιχεία πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουν ε, παλιά, ε, παλιές νοοτροπίες ε, και έθιμα καθώς και η εφαρμογή της νοοτροπίας της κάστας. Θα πρέπει όμως ε, η Μαυριτανία να διορθώσει αυτή την αποτρόπαια κατάσταση και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πρέντα που ήταν ο πρωτεργάτης του ψηφίσματός μας που είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκασμπάρα δεν τον βλέπω στην αίθουσα, οπότε δίνω το λόγο στην κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τι περίεργη χώρα η Μαυρετανία. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Μέρμερτ Χούλαμπετ Χασή, πρόεδρος της Μαυρετανία, με στρατηγικό πραξικόπημα ε, ανέτρεψε τον πρώτο πραγματικά δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο μετά την ε, ανεξαρτησία. Ε, ε, ε, ωστόσο εμείς χαϊδεύουμε τη χώρα αυτή γιατί έδιωξε την ακμή αλλά παρόλα αυτά αποτελεί κέντρο διακίνησης ναρκωτικών και οπωσδήποτε κέντρο θεσμοθετημένου ρατσισμού και δουλείας. Παρά την κατάργηση του 81 και την ποινικοποίηση το 2007 της δουλείας αυτή εξακολουθεί να υπάρχει από το 2008 ε, ο Μπιράμ Νταν Αμπέιντε, γιος ελευθερωμένων σκλάβων Χαρατσίν, ε, βρίσκεται στη φυλακή ε, γιατί παλεύει για τα δικαιώματα πίσω από κάποιες θρησκευτικές υποτίθεται αιτιάσεις βρίσκεται ακόμα στη φυλακή και κινδυνεύει τη θανατική ποινή. Για όλους αυτούς τους λόγους θα υπερψηφίζω. Ευχαριστώ πολύ. Καστάλντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μία ακόμα φορά μιλάμε εδώ για τον Μπιράμ Ντάμα Χαμπέιτ, έναν ε, φυλακισμένο και βασανισμένο θαραλέο ε, ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσπαθεί να ε, σώσει τον κόσμο από μία πληγή αυτήν της δουλείας. Η δουλεία ήδη έχει καταργηθεί επισήμως από το 1981 αλλά εξακολουθεί να είναι συστημικά ενταγμένη στην χώρα αυτή περισσότερες από 200 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί στην χώρα αυτή ε, άμεσα αλλά και άλλες χρηματοδοτήσεις ε, μέσω άλλων ταμείων ε, έτσι ώστε να βοηθηθεί η χώρα αυτή αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία κοτονού πραγματική χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι δυνατόν να κλείνει τα μάτια η Ευρώπη γιατί διαφορετικά θα γίνει και αυτή συνένοχη ε, σε αυτό το καθεστώς το οποίο έχει καταδικάσει και φυλακίσει έναν άνθρωπο σύμβολο του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Μπιράμ Ντάχα Αμπέιτ πρέπει να αποφυλακιστεί αμέσως. Θα πρέπει να ελευθερωθεί μαζί με ολόκληρο το λαό της Μαυριτανίας. Ο κύριος Επιτίδιος. Είναι ίσως απίστευτο, αλλά στον 21ο αιώνα περισσότερο από το 20% του πληθυσμού ε, της Μαυριτανίας είναι σκλάβοι. η, κυβέρνηση της χώρας αντί να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την απαράδεκτη αυτή κατάσταση έκανε κάτι απλό συνέλαβε τον κύριο αμπέιντ πρόεδρο μιας ακτιβιστικής οργανώσεως ε, κατά της δουλείας με ανυπόστατες κατηγορίες καθώς επίσης και ορισμένα από τα στελέχη της οργανώσεώς του. θα μου πείτε ότι η στάση της κυβερνήσεως της μαυριτανίας ενδεχομένως να μην προκαλεί έκπληξη διότι είναι αντιδημοκρατική και θα την καταδικάσουμε. όταν όμως την ίδια στάση τηρεί και μια κυβέρνηση δημοκρατικής χώρας όπως η κυβέρνηση της ελλάδος η οποία κατόπιν ομής παρεμβάσεως του πρωθυπουργού στη δικαιοσύνη κρατά επί 14 μήνες παράνομα στη φυλακή τον αρχηγό βουλευτές και στελέχη του τρίτου σε δύναμη πολιτικού κόμματος της ελλάδος της χρυσής αυγής γιατί δεν δείχνουμε την ίδια ευαισθησία. το θέμα το γνωρίζετε γιατί έχουν αναφερθεί σε αυτό κατ' επανάληψη και άλλοι δύο συναδελφοί μου ευρωβουλευτές. το αναφέρω όμως για να δείξω πόση υποκρισία υπάρχει σε αυτή την αίθουσα. εάν πιστεύετε ότι έχω άδικο και σα αδικό παρακαλώ με τη συμπεριφορά σα να με διαψεύσετε. Ευχαριστώ. Ο Βέντα. Ε, Κύριε Πρόεδρε, η δουλεία καταργήθηκε στη Μαυριτανία το 1981, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν διατάξεις που να εφαρμόζουν την ποινικοποίηση. Και δυστυχώ είναι κληρονομική η δουλεία και περιορίζεται κυρίως σε μία εθνοτική ομάδα, τους Χαρατίν. Και μάλιστα κυρίω σε μια εθνοτικη ομαδα του χαρατιν και μαλιστα δεν μπορουμε να ανεχτουμε τις παραβιάσει ανθρωπινων δικαιωματων γιατι λαμβανουν χωρα σε μια χωρα σαν τη Μευρετανία που συμμετέχει στι χώρε ΑΚΕ. Θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Χρειάζεται φυσικά η δράση των τοπικών ε, ακτιβιστών. Γι' αυτό στηρίζουμε ιδιαίτερα τι δράσει του κυρίου Μπιράμ Νταχαμπέιτ και άλλων ακτιβιστών που φυλακίστηκαν για τη δράση του. Ζητούμε αποφυλάκηση του Πειράμα Μπέιτ και άλλων ε, ακτιβιστών, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα της δουλείας στη Μαυριτανία. Κάποιες δημοκρατικές ενέργειες και ενέργειες υπέρ της σταθερότητας, ε, μόνο έτσι θα, θα βελτιωθούν οι σχέσεις ε, Μαυριτανίας και Ευρωπαϊκή Ένωσης και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας αυτής. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Κύριε Πρόεδρε, Πρόκειται για την τρίτη χρονιά κατά την οποία συζητάμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μιλάμε για τη δουλεία στη σημερινή εποχή αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η Μαυριτανία ήταν η τελευταία χώρα η οποία επίσημα υποτίθεται κατάργησε τη δουλεία. Όμως μετά από τρία χρόνια πολλοί πιστεύουν ότι μέχρι και 20% περίπου του πληθυσμού εξακολουθούν να ζουν αυτό λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να το δεχτούμε, να καλέσουμε τη Μαυριτανία να εφαρμόζει τους ε, κανόνες της χώρας και να δώσουμε την ευκαιρία στους σκλάβους ε, να γίνουν κυρίαρχοι της γης τους. Ε, επίσης οφείλουμε να απελευθερωθεί ο, ο κ. Ταπέτ γιατί πραγματικά βρίσκεται παράνομα στη φυλακή. Περνάμε στο Catch the και πάλι έχουμε πολλούς συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Γκέριγκερ, δεν μπορούμε δυστυχώς να ικανοποιήσουμε όλους όσους ζήτησαν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Μπιράμ Ταχαμπέιντ είναι ακτιβιστής και το 2013 για τη δράση του έλαβε το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Δυστυχώς ε, τον ε, Νοέμβριο μαζί με πολλούς ακτιβιστές ε, ο Μπιράμ Μπέιντ και σε μια ειρηνική διαδήλωση για την κατάρριξη της δουλείας συνελήθη και φυλακίστηκε. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή του. Η Μαυριτανία είναι εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της συμφωνίας με τις χώρες ΑΚΕ. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά της δουλείας ε, και οποιασδήποτε, οποιοδήποτε άλλο περιορισμού της ανθρώπινης ελευθερίας. Ε, ζητούμε από την κυβέρνηση της ε, Μαυριτανίας να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις και να θεσπίσει τις κατάλληλες νομοθετικές διατάξεις για να υπερασπίσει τους πολίτες της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΕΔ θα πρέπει να συσφίξουν τις σχέσεις με την ε, Μαυριτανία υπογραμμίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης ε, κάθε μορφής εξανδραποδισμού και φυσικά προστασίας των ακτιβιστών. Ο κύριος Μαριάς. Πράγματι εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν ψήφισμα που αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες όπως ήταν το προηγούμενο ψήφισμα που αφορούσε τη Βενεζουέλα η δουλεία είναι γενικευμένο καθεστώς στη μαυριτανία και πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις κατά των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του μπιράμ νταχ αμπέι. καταδικάζω λοιπόν τη δουλεία που υπάρχει στη μαυριτανία υποστηρίζω το ψήφισμα και ορθώς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ασχολείται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. οφείλει όμως να κάνει το ίδιο και για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ίδια την ευρωπαϊκή ένωση στις χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό μνημόνιο στις χώρες όπου η τρόικα παραβιάζει βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα φτάσαμε σε σημείο η επιτροπή να πει απαντώντας σε ερώτηση ότι δεν μπορεί να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίπτωση της ελλάδος διότι εκεί εφαρμόζεται το μνημόνιο. είναι απαράδεκτο και το καταδικάζουμε. <coughs> Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συζητούμε για μια χώρα που είναι παλιός εταίρος μας ε, και που δυστυχώς εφαρμόζει εμπράκτο στη δουλεία. Η Μαυριτανία, κυρίες και κύριοι, είναι μέλος της Ευρωμεσογειακής Ένωσης. Είναι μέλος ε, μιας ένωσης που ξεκινήσαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την θερμή μου συμπαράσταση και στήριξη του ψηφίσματος. Και περιμένω από την ύπατη εκπρόσωπο, την κυρία Μογκερίνη, να κάνει ό,τι μπορεί για να απελευθερωθεί ο κύριος Μπιράμ Ταχαμπέιντ, να αποφυλακιστεί, γιατί είναι σύμβολο του αγώνα κατά ενός συστήματος και κυρίως κατά των απάνθρωπων συνθήκων στο οποίο διαβεί μεγάλο ποσοστό του μαυριτανικού ε, Θα ήθελα να ενθαρρύνω λοιπόν την κυρία Μογκερίνη για να αναλάβει άμεση δράση. Ευχαριστώ. Grazie signor Presidente, onorevole. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας πω με πολύ μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε αυτή την, ε, το ψήφισμα καταπήγοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μαυρτανία, κυρίως για την περίπτωση του Μπιράμ Νταλαμπέιτ αφορά το ψήφισμα και άλλα μέλη της οργάνωσής του της ΙΡΑ. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την περίπτωση του Μπιράμ, ο οποίος είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Μαυριτανία, ακτιβιστής ε, κατά της δουλείας, έχει καταδικαστεί πολλές φορές και κατηγορείται για αποστασία προδοσία το 2012. Θεωρώ ότι ε, ο ίδιος είναι εκείνο που αναζωγόνησε το κίνημα κατά της ε, δουλείας. Ε, είναι εκείνο που είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως πολιτικός όν και ως ήταν επίσης υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές. Ο Μπιράμ συνελήφθη από κοινού με άλλα μέλη της οργάνωσής του στο πλαίσιο μιας περιπολίας, μιας επίθεσης παράνομης και αυτό έγινε ε, μόνο και μόνο επειδή ήταν μέλλον αυτής της οργάνωσης. Ε, υπήρξαν ε, καταγγελίες ότι δεν σέβεται τα βασικά δικαιώματα των Μαυριτανών ε, στη Μαυρτανία βεβαίως ε, ζουν πάρα πολλοί μαύροι καθότι ε, γειτονεύει με τη Σενεγάλη. Οι αρχές της Μαυρτανίας δηλώνουν ότι τώρα ο Μπιράμ βρίσκεται στα χέρια των δικαστών και θα περιμένει τη δικαστική διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις συλλήψεις. Μέσα από την οργάνωση της Μαυρτανίας που έχουμε και εμείς είμαστε σε συνεχή επαφή με την οργάνωση του Μπιράμ. Ενημερωνόμαστε για την κατάστασή του στη φυλακή, για το πώς διεξάγεται, πώς προχωράνε τα πράγματα, κυρίως σε δικαστικό επίπεδο. Πρέπει να δράξουμε κάθε ευκαιρία για να έχουμε διάλογο με τις αρμόδιες αρχές. Οι πρέσβεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση του Μπιράμ ε, ενημερώθηκαν από τον Πρωθυπουργό μέσα μετά τη σύλληψή του. Επίσης έγιναν και άλλες συζητήσεις 15 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που προβλέπεται από τη Συμφωνία της Κοτονού. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του Μπιράν. Και επίση ανέφερε ότι δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση για καμία εθνοτική μειονότητα. Αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο για την ενότητα και τη σταθερότητα τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ τη σύνεγγυ την περίπτωση του Μπιράν Νταλαμπέιτ. Επίση θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε διάλογο με τι αρμόδιε αρχέ, με την κοινωνία των πολιτών για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δίκαιη δίκη. Όπω και αν εξελιχθεί η κατάσταση, εμεί δεν θα διστάσουμε μπορούμε να παρέμβουμε αν χρειαστεί. Ενημερωθήκαμε ότι η δίκη τελικά ίσως αρχίσει και σήμερα μάλιστα και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται επί τόπου παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ τη δίκη, η οποία δίκη μέσα εδώ πρέπει να λάβει χώρα το στομότερο δυνατόν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τον τακτικό διάλογο με τη Μαυριτανία για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα στηρίζουμε την κυβέρνηση και τη δέσμευσή της να ενισχύσει τις ε, αρμόδιες αρχές και επίσης να θεσπίσει ε, νομοθετικά διατάγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνει ακόμα περισσότερα. Ε, τον Μάρτιο του 2014 η Μαυριτανία κατέθεσε χαρτιπορία στα Ηνωμένα Έθνη με μια σειρά συστάσεων για να εξαλειφθεί η δουλεία ακόμα και τελευταία της μορφή. Επίσης συμφωνήθηκε να υπάρχει ένα ειδικό ποινικό δικαστήριο που θα ασχολείται με περιπτώσεις δουλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την κυβέρνηση να προχωρήσει με αυτό το χάρτη πορεία. Και εδώ είμαστε σε στενή επαφή με το αρμόδιο οργανισμό των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης έχουμε και περιοδικέ επαφές με τους αμήντορε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. μα δίνουν έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα τη κατάσταση για να κατανοήσουμε και τι γίνεται και σε επίπεδο κυβέρνηση. Εδώ θέλουμε να επενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μάλιστα τρία προγράμματα ε, στο πλαίσιο ε, τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τρία προγράμματα που θα ε, βοηθήσουν τις ΜΚΟ. Ε, όμως αυτή εδώ η περίπτωση που έχουμε μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σημειωθεί και άλλη πρόοδος και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι στο πλαίσιο του διαλόγου ε, και της συνεργασίας με τη Μαυριτανία το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα προβλήματα της δουλείας θα θυγούν η περίπτωση του Μπιράμντα Αμπέιτ αλλά και άλλες περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον θα παραμείνουν για μας πρώτο θέμα της μερίσιας διάταξης. Θα συνεχίσουν να είναι προτεραιότητές μας και στο πλαίσιο των διπλωματικών μας δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Ταλαβέντοβα. Ρογαρία, Λίγη ησυχία παρακαλώ. Γιατί είναι αδύνατο να ακούσουμε τους ομιλητές με φασαρία στην αίθουσα. Θέρμο παρακαλώ λοιπόν ησυχία. Περνάμε στο επόμενο σημείο.